ιδιαίτερα Ουκρανία και Λευκορωσία. Έχει και διδακτορικό ε, στην ιστορία στην πολιτική, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών και θα μιλήσει για την ε, καλή διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Παρακαλώ κύριε Αντάμσκι, έχετε το λόγο. Με μικρόφωνο, παρακαλούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, στα γερμανικά, κυρίες και κύριοι. Στα αγγλικά τώρα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ευκαιρία που έχω να μοιραστώ με ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο τις ε, προσωπικές μου απόψεις για την Ανατολική ε, Γειτονία και την πρώτη πλατφόρμα για τη δημοκρατία, σταθερότητα και το κράτος δικαίου ιδιαίτερος. Ε, Χωρίς καμιά αμφιβολία η ανατολική γειτονία και η εταιρική σχέση είναι μια καλή ε, πρωτοβουλία για να ε, διατηρηθούν ε, τα ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Γειτονία, να υπάρξει και χρηματοδότηση και υποστήριξη των ανατολικών μας εταίρων. Η Ανατολική Γειτονία διευκολύνει βέβαια και τις επαφές μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών και των ηγετών των κρατών αυτών. Και είναι μάλλον το καλύτερο μέσο που θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν ε, δεχτεί επικρίσεις. Από την άλλη όμως η Ανατολική Γειτονία προσφέρει πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις τεράστιες προσδοκίες που έχει γεννήσει και τις ελπίδες των κοινωνιών αυτών των κρατών, κυρίως επειδή είναι ισχνά και πενιχρά τα οικονομικά, γιατί δεν υπάρχει η βούληση, η πολιτική, δεν υπάρχει δυνατότητα για την ε, πρόταση κάποιων λύσεων που θα ήταν επιθυμητές για ε, τις χώρες αυτές και από πλευρά των ανατολικών εταίρων και των κοινωνιών τους βλέπε διευκόλυνση ε, και άρση της υποχρέωσης ε, θεώρησης διαβατηρίων. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πει κανείς ότι στην Ουκρανία, τη χώρα ε, που ζω 10 μέρες το μήνα, κανείς δεν γνώριζε αυτά τα θέματα με εξαίρεση κάποιους εμπειρογνώμονες ή πολιτικούς. Ουδής γνωρίζει την Ουκρανία τι εστί ατολική εταιρική σχέση πολύ περισσότερο οι πολίτες και η πολιτική ελίτ πολύ συχνά γνωρίζουν ελάχιστα ε, για τον ε, χώρο ελευθέρων συναλλαγών, για να μην μιλήσω και για άλλα στοιχεία της κοινωτικής πολιτικής. Ε, ο σημαντικότερος λόγος όμως, για ποιο λόγο δεν υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος, είναι πολύ περιορισμένος, είναι η εσωτερική κατάσταση στις χώρες αυτές της Ανατολικής Γειτονίας. Πέντε χρόνια έχουμε αυτό το μέσο της Ανατολικής Γειτονίας. Και χώρες αυτές ούτε περισσότερο δημοκρατικές έχουν γίνει, ούτε πιο σταθερές. Ακόμα και εκείνες που θέλουν να, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Μολδαβία, η Γεωργία, η Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει ε, κάνει μεταρρυθμίσεις βέβαια στη διοίκηση και στην οικονομία, αλλά όχι στη ε, δημοκρατία, ούτε υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες ε, για να περιοριστεί η τεράστια διαφθορά και να επέλθει ένα κράτος δικαίου. Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου, η σημερινή κατάσταση ήταν προβλέψιμη και δεν θα πρέπει να θεωρείται έκπληξη ούτε ε, λόγος για αδράνεια ή για απελπισία. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι η ανατολική γειτονία μπορεί να ε, επιτύχει μόνο εφόσον οι χώρες ε, της γειτονίας διαθετήσουν ε, το κράτος δικαίου και βελτιώσουν την καλή διακυβέρνησή τους. Και κυρίως να περιορίσουν τη διαφθορά. Δεν είναι προϋπόθεση η δημοκρατία για τις μεταρρυθμίσεις, το αντίθετο ισχύει. Χρηματοδοτικά έχουμε μόνο δύο μέσα στη διάθεσή μας στην Ένωση για να ε, οθήσουμε τις χώρες αυτές να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Πρώτον, Υπάρχει ένας ε, βαθύς και ευρύς χώρος ελευθέρων συναλλαγών. Όσο ε, πιο σύντομα εφαρμοστεί και υλοποιηθεί, τόσο θα βελτιώσει την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών. Και αυτό με κάνει να προτείνω το εξής η εφαρμογή αυτού του χώρου ελευθέρων συναλλαγών θα φέρει πολύ περισσότερα και για τη δημοκρατία και για το κράτος δικαίου από την αιρεσιμότητα ε, από το να ήταν μέσω πίεσης για να βγει από τη φυλακή η κυρία Τιμοσέγκο ε, ή ε, για να εγκριθούν κάποιοι νόμοι κατά των διακρίσεων. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει ως όθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν η ε, άση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο βήμα που να διευκολύνει τόσο πολύ τη ε, μεγάλη μεταφορά των κοινοτικών νοοτροπιών, πρακτικών κτλ. από την ε, απρόσκοπτη διεξαγωγή των μετακινήσεων και των ταξιδιών χωρίς θεώρηση διαβατηρίων. Τι εννοώ η Βίζα δεν προστατεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από το έγκλημα ούτε από τους παράνομους ε, μετανάστες και ε, εργαζόμενους. Εμποδίζει περισσότερο τους τουρίστες και τους φοιτητές που θέλουν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά κάποια εγκληματικά στοιχεία. Δεν προστατεύει ας πούμε, το μικρό λαθεμπόριο και ε, τις παρανομίες. Αυτοί ξέρουν πώς να παρακάμπτουν τη Βίζα. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες, πολυμερείς, ε, θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε, αλλά όπως σας είπα ήδη, ε, οι δράσεις, τα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μικρή ε, επιρροή και μικρή ορατότητα. Με εξαίρεση τις διασκέψεις. Υπάρχουν διάφορες διασκέψεις και διοργανώσεις για την Ανατολική Γειτονία, αλλά κατά την άποψή μου Δύο είναι τα μεγάλα εμπόδια σε αυτή την υπόθεση. Και καλύτερα θα είναι να επικεντρωθούμε στον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών, στον εξυγχρονισμό των χωρών, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, παράδειγμα την Ουκρανία, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, αυτό ε, που ε, ισχύει για τις μίζες είναι πολύ διαφορετική κατάσταση σε σχέση με τα όσα ισχύουν στην Ουκρανία. Δηλαδή, στις χώρες ανατολικής γειτονίας χρειάζεται κανείς να δωροδοκίσει ένα υπάλληλο για να κάνει τη δουλειά του. Εκεί θα πρέπει να χτυπηθεί αυτό το κακό στη ρίζα του και το κράτος δικαίου είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση στην Ανατολική Ευρώπη. Ένα τελευταίο. Να πω δύο λόγια για τη Ρωσία. Όπως είπε ο Πρόεδρος, εργάζομαι στο κέντρο πολωνο-ρωσικού διαλόγου και κατανόησης. Πριν από μία διετία συνέταξα μαζί με κάποιους άλλους μία έκθεση που απεικονίζει και προτείνει δυνατότητες συνεργασίας της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ανατολικής Γειτονίας. Ε, τι ενδιαφέρον είχε αυτή η έκθεση. Συμμετείχαν και πολλοί Ρώσοι ε, ε, εμπειρογνώμονες και από πανεπιστήμια της Ρωσίας ο τελικός στόχος μας θα, ε, πρέπει να είναι η ένταξη της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και να έρθει όσο γίνεται πιο κοντά η ρωσική νομοθεσία στο κοινοτικό και εκτιμένο. Μπορεί ας πούμε να έχει ένα καθεστώς αντίστοιχο της Νορβηγίας ή της Ελβετίας τελικά ε, στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ρωσία. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Ρωσία ασκεί τεράστιες πιέσεις στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας που ε, επιθυμούν να υπογράψουν αυτές τις ενισχυμένες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πίεση λοιπόν που δεν χαλαρώνει για να μην υπογράψουν Κατά την άποψή μου δεν αποδίδει αυτή η πολιτική, δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και δεν επιτυχάνει το στόχο της. Πιθανότατα οι Ρώσοι πολιτικοί που ασκούν αυτές τις πιέσεις μπορούν να θεωρηθούν μέχρι και ιδρυτές πατέρες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των κρατών αυτών, γιατί τους πρόχνουν προς την κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, ε, η Ρωσία τους κατηγορεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τους προστατεύουν. Ε, θα πρέπει να δούμε εμείς όμως πώς θα φέρουμε πιο κοντά τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα πείσουμε τη Ρωσία να συνεργάζεται σύμφωνα με τις βέλτιστες κοινοτικές πρακτικές και το κοινοτικό κεκτημένο. Στην έκθεσή μας ε, πριν από δύο χρόνια προτείνουμε κάποια ε, θέματα σχετικά και πώς θα φέρουμε πιο κοντά τη Ρωσία. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες σας. Μας δίνουν πολύ τροφή για σκέψη. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Σουτέλα να λάβει το λόγο. Θα μιλήσει για οικονομία σε μετάβαση και κυρίως τις προοπτικές σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για επισκέπτη καθηγητή στο Παρίσι, στη Σχολή Ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Έχει διατελέσει ε, τόσο στην Φιλανδία όσο και στη Ρωσία έχει ασχοληθεί με θέματα του ευρωπαϊκού χώρου. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Ως οικονομολόγος θα μιλήσω εν συντομία για κίνητρα, οικονομία και ανάπτυξη. Τα κίνητρα, όπως γνωρίζουμε, τα κίνητρα που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των προοπτικών προσχώρησης στη, στο ΝΑΤΟ, τον ΩΣΑ και το καθεξής ήταν πολύ σημαντικά για την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και άλλων για τις χώρες αυτές σε μετάβαση, τις οικονομίες όπως ονομάζουμε σε μετάβαση, ε, για όσους βεβαίως είχαν ρεαλιστικές προοπτικές για ένταξη σε αυτούς τους οργανισμούς ήταν πάντα πολύ πιο αδύναμες, ε, αδύναμα τα επιχειρήματα για την παροχή κινήτρων σε εκείνα τα κράτη τα οποία για το ορατό τουλάχιστον μέλλον δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιθανά ε, μέλη ή μελλοντικά μέλη. Κράτη τα οποία θέλουν, ε, στους οργανισμούς που ε, ήθελα να ταχθούν τα κράτη αυτά και που το ευρωπαϊκή σήμερα. Η, τα κίνητρα λοιπόν μπορούν να προσφέρονται. Είναι στην περίπτωση αυτή σχετικά περιορισμένα και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από τις χώρες εταίρους πολλές είναι αυτές οι οποίες έχουν εξειδικευτεί στην ανάληψη δεσμεύσεων τα τελευταία χρόνια. Στα διάφορα μέσα και προγράμματα με κίνητρα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι τα κίνητρα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Και θα αναφερθώ στην οικονομική ανάπτυξη και τη σύγχρονη θεωρία οικονομικής ανάπτυξης ως καθηγητής στο παρελθόν και στο παρόν. Ξέρετε, η σοφία ξεκινάει όταν κανείς ε, μπορεί να διαχωρίσει μεταξύ δύο ειδών οικονομίας, αυτών που λειτουργούν ικανοποιητικά, ο ΩΣΑ δηλαδή, χωρίς του ΩΣΑ, και αυτών που είναι αναποτελεσματικές και εξασφαλίζουν σχετικά χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων και ευημερία για τους πολίτες τους και εν γέννη έχουν τέτοια αδυναμία. Οι αποτελεσματικές οικονομίες ε, αναπτύσσονται με την καινοτομία, η οποία ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί, δάπανα, ε, είναι πολύ δάπανη, πολλές φορές αποτυγχάνει. Άρα η ανάπτυξη αυτών των αποτελεσματικών οικονομιών είναι βραδία πάντα. Ενώ οι μη αποτελεσματικές οικονομίες μπορούν να λειτουργούν, να αναπτύσσονται γρήγορα εφόσον μπορούν να προσαρμόζονται με καλύτερα βασικά αγαθά, ε, τεχνολογία, θεσμούς, ε, όλα αυτά τα οποία έχουν εφεύρει και δοκιμάσει στην ε, πράξη κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κορέα στο παρελθόν αναπτύχθηκαν γρήγορα, γι' αυτό χώρες όπως η Κίνα στο παρόν αναπτύσσεται γρήγορα και γι' αυτό αναπτύσσονται γρήγορα ή θα αναπτύσσονται μάλλον γρήγορα στο μέλλον χώρες ε, της Αφρικής. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της ε, ανάπτυξης που στηρίζεται στην καινοτομία ή της ανάπτυξης που στηρίζεται στην απομίμηση, αν θέλετε, στην ε, παρακολούθηση της καινοτομίας κάποιων άλλων, για να είμαι πιο ευγενικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε όχι το γιατί, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα, εάν όπως ιστορικά είδαμε την Κίνα, την ε, Ινδία και τη Ρωσία ακόμα, ε, σε θέση να αναπτυχθούν γρήγορα ή να παρακολουθήσουν την ε, καινοτομία άλλων, να απομιμηθούν. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ή η αδυναμία της παρακολούθησης αυτών των ρυθμών μπορεί να οφείλεται σε πολιτική αβεβαιότητα, ακόμη και σε εμφυλίους πολέμους ή, όπως δείχνει και η έρευνα, σε λόγους βαθιά ριζωμένους και ιστορικούς. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ λεπτό θέμα την ε, διάκριση δηλαδή μεταξύ προκαταλήψεων και γνώσεων που μπορεί να κρίνουν το κατά πόσο μπορεί μια χώρα να εισαγάγει καινοτόμες μεθόδους. Ίσως όμως να μην είναι δυνατόν για όλες τις χώρες που θα θέλαμε να μπορούν να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη να το πράξουν σε ιδεώδεις συνθήκες. Επίσης, πολύ σημαντικό και άμεσης ε, σημασίας για την ε, συνεδρίασή σας είναι το ότι οι θεσμικές δομές, οι κατάλληλες για μια οικονομία στηριζόμενη στην καινοτομία, με ανάπτυξη, στηριζόμενη στην οικονομία, μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές μιας βάσεως οικονομίας παρακολούθησης της καινοτομίας. Πράγμα το οποίο είναι και το κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί όταν χορηγούμε κίνητρα σε οικονομίες που θέλουμε να οθήσουμε, να εξωθήσουμε στην παρακολούθηση και κάλυψη του χαμένου εδάφου στην καινοτομία. Και γιατί το θέλουμε αυτό, για ένα πολύ απλό ε, λόγο, ότι η ανάπτυξη της όλης οικονομίας είναι το σύνολο είναι το άθροισμα της οικονομίας που στηρίζεται στην καινοτομία και των οικονομιών των χωρών που παρακολουθούν την ε, καινοτομία των άλλων. Και άρα όσο πιο γρήγορα προχωρούν οι δεύτερες χώρες, η ομάδα των δεύτερων χωρών, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται και η συνολική οικονομία, η παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα στο να αντιληφθούμε ότι η πρόσβαση στην αγορά και η κινητικότητα είναι ζητήματα κλειδιά, είναι ζητήματα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε, να υποσχεθούμε ως ε, κίνητρα και εκείνους τους ε, γείτονές μας που θέλουμε να οθήσουμε στην κάλυψη του χαμένου εδάφους και την παρακολούθηση της κοινοτομίας. Και έτσι όσο παράξενο και να το βλέπω αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολιτικά, πολιτική επιλογή του να στηρίζουμε κάποιες χώρες ε, όταν μας απασχολεί ένας ενδεχόμενος κίνδυνος σχετικός με την πρόσβαση σε αγορές ή αν τελικά ένας από τους γίνατονες ε, έχει πολύ, μικρή, πολύ μικρά μεγέθη παροχής υπηρεσιών στις αγορές μας. Η κινητικότητα για προφανείς λόγους που εξέθεσε άλλωστε ο προλαλής σας, η κινητικότητα των φοιτητών και των επαγγελματιών φυσικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την παροχή κινήτρων για την θεσμική και κανονιστική προσέγγιση. Καταρχάς, διότι η ελκυστικότητα, η αξιοπιστία της Ένωσης είναι πολύ μικρότερη από όταν πριν από 20 χρόνια, πρώτον. Δεύτερον, διότι και για λόγους ιστορικούς και για λόγους οικονομικής λογικής, δηλαδή επειδή οι θεσμοί είναι διαφορετικοί στην, ε, στην ομάδα των κρατών της καινοτομία και εκείνων που παρακολουθούν την καινοτομία, δεν μπορούμε να ε, προσφέρουμε τις ίδιες λύσεις ε, στους εταίρους ή γείτονέ μας, με αυτές που είχαμε στις δικές μας οικονομίες αξιοποιήσει επιτυχώς. ξέρω ότι αυτό είναι περίπλοκο, αλλά θα ήθελα να το αξιοποιήσουμε ως ένα σημείο κίνησης και κυρίως καθώς οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Και η υπαγωγή σε και όρους δεν φέρνει συχνά αποτελέσματα συχνά δεν φέρνει αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κυριαλιστές ως προς την ε, προσδοκία της υλοποίηση των όρων και προϋποθέσεων. Για δε, τις, ε, για δε λόγους ε, κινήτρων δεν νομίζω ότι η επιβολή όλο και περισσότερων όρων μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ε, τα κίνητρα αλλά και η αντίστροφη μορφή, ε, τα, οι κυρώσεις δηλαδή, μπορεί να φέρουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στιούαρτ είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος ε, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια ε, ε, του Βερολίνου. Θα βασιστώ σε δύο ε, πτυχές της πολυμερούς σχέσης αυτής. Θα μιλήσω για την τέταρτη πλατφόρμα σε σχέση με τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων της κοινωνίας από την κοινωνία των πολιτών και θα μιλήσω και για το ρόλο της ε, κοινωνίας ε, των ε, πολιτών μέσα στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Όσο αφορά τις επαφές μεταξύ ανθρώπων, έχω ασχοληθεί με θέματα εκπαίδευσης, νεότητας, πολιτισμού και καινοτομίας. Οι στόχοι αυτής της πλατφόρμας, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αφορούν μέσα ε, τα οποία είναι και τα πλέον κατάλληλα. Θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις περισσότερο, κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ σύμφωνα και με τον τίτλο της ημερίδας. Ο μόνος τρόπος για να μετρήσουμε την, ε, τις επιπτώσεις, ο μόνος τρόπος είναι καθαρά ποσοτικός. Η εκτίμηση είναι θετική διότι είδαμε σε όλους τομείς ότι από το 2009 με την εκκίνηση της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης γίνεται μία συνεχής χρηματοδότηση αυτών των ε, τομέων που ολοένα και διονγκούται. Υπάρχει λοιπόν η χρηματική αρρωγή και μία ανωδική τάση χρηματοδότησης. Πέρα όμως από μία τέτοια εκτίμηση, όταν θέλουμε να κρίνουμε την τέταρτη πλατφόρμα και την πολυμερή αυτή συνεργασία, θα πρέπει να σταθούμε και σε άλλες παραμέτρους, διότι η φύση αυτής της πλατφόρμας αφορά μεμονωμένες εμπειρίες. Άρα τα παράγωγα αυτής της ε, πλατφόρμας είναι πολλές φορές ε, σχετικά άειλα θα μπορούσα να πω και αφορούν μία μορφή διάδρασης. Μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πέντε τρόπους για να προωθήσουμε τη δυναμική αυτής της πλατφόρμας και των επαφών. Πρώτον, και σε σχέση με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχία των επαφών αφορά την κινητικότητα και την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Άρα αυτή η ατζέντα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων αφορά τους προσανατολάς εταίρους και τις σχετικές επαφές και τις οποίες εμβαθύνουμε. Είναι μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να προβούμε σε μία στοχοθέτηση, δηλαδή να μιλήσουμε για μη κυβερνητικό και μη γραφειοκρατικό επίπεδο. Αν δείτε τι έχει γίνει στον τομέα του πολιτισμού, βλέπετε ότι μιλάμε για πολιτισμικές πολιτικές και τη σχετική διοικητική τους πλαισίωση. Εάν αυτός ο τομέας είναι επιτυχής, δεν πρέπει να τον ε, εγκαταλείψουμε. Αυτή η πλατφόρμα όμως θέλει να εξεύρει ε, τρόπους συνεργασίας εκτός κυβερνητικού πλαισίου. Σε σχέση με την νεότητα, πρόκειται για σημαντική κατηγορία επίσης, διότι οι πολίτες ε, των χωρών της ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης θα πρέπει να αφορούν επαφές από πολύ νεαρή ηλικία μέσα στα πλαίσια μιας καθημερινότητας για να αυξήσουμε και τις γνώσεις, ιδιαίτερα την ε, εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σε νεαρή ηλικία είναι πολύ πιο εύκολο να αρχίσουμε με παρόμοιες επαφές. Τέταρτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτά τα σχήματα διάδοσης, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τις ευκαιρίες που διανοίγονται από την τέταρτη αυτή πλατφόρμα. Η ανατολική εταιρική σχέση δεν είναι τόσο ευρέως γνωστή στους πολίτες ως προς τις ευκαιρίες που διανοίγει και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι εταίροι που συμμετέχουν με υποτροφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής συνεισφέρουν. Δηλαδή δεν φεύγουν με γνώσεις, αλλά μπορούν να προωθήσουν την καινοτόμο γνώση για τη ζωή σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή πρόκειται για μία αμφίδρομη πορεία. Ως προς τη δεύτερη πτυχή, δηλαδή το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την ε, πολυμερή σχέση αυτής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία των πολιτών ε, ε, δρά άμεσα και πολύ περισσότερο από την εκκίνηση του προγράμματος και μετά. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη τα φόρα των, ε, της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν ενεργά. Μιλάμε για εθνικές ε, πλατφόρμες και θεματικές εργασίες μέσα στα πλαίσια της ε, πολυμερούς αυτής συνεργασίας. Και επίσης έχει δημιουργηθεί πρόσφατα μια πέμπτη πλατφόρμα για τον κοινωνικό διάλογο που αποτελεί ε, σοβαρή και πρόσφατη εξέλιξη διότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια αναγκαία προστίκη του σχήματος αυτού συνεργασίας. Ο ρόλος της κοινωνίας ε, των πολιτών θεσμοθετεί τέλο ένα και περισσότερο. Υπάρχει μια γραμματεία εδώ στις ε, Βρυξέλλες δεν είναι μία ad hoc μορφή συνεργασίας, αλλά μία θεσμοθετημένη μορφή μέσα σε κυβερνητικά πλαίσια. Αν δούμε τις ε, επιπτώσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά ευεργετικά βήματα, διότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσα στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης και υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση ε, έτσι ώστε να, να υπάρχει αυτή η ανάδραση από την κοινωνία των πολιτών. Επίσης βοηθούμε τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε μια κοινή ατζέντα μέσα στα πλαίσια μιας επαγγελματικής προσέγγισης. Επίσης η κοινωνία των πολιτών βοήθησε ιδιαίτερα τη Λευκορωσία διότι η Λευκορωσία ασχολείται με το πολυμερές αυτό πλαίσιο και η κοινωνία των πολιτών ήταν πολύ δραστήρια από πλευράς ε, Λευκορωσίας. Όμως υπήρξαν λιγότερες επιπτώσεις ως προς την επιρροή της ε, κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια της ανατολικής συνεργασίας συμμετέχει ευρύτερα σε όλα αυτά τα φόρα, όμως ελοχεύουν και ορισμένοι κίνδυνοι. Άλλες, ε, άλλες ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεν είναι τόσο κοντά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλείονται. Δεν υπάρχει πάντα πλουραλισμός ε, δραστηριοτήτων και το φόρουμ αυτό της κοινωνίας ε, των πολιτών μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικό ε, ότι διέπει όλες, όλη την κοινωνία των πολιτών, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Και επίσης ελοχεύει ο κίνδυνος αυτό το φόρουμ να ε, διονγκώνει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, αντιπρο... και της αντιπροσώπευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει να είναι ένας ε, διαμεσολαβητής, ο οποίος να μας δίνει και αυτό το feedback όταν το χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία ευελιξία και στα πλαίσια αυτού του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και τις ε, σχετικές οργανώσεις και μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής της κοινωνίας των ε, πολιτών από τις πολυμερείς ε, πλατφόρμες. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε το ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας την προσοχή στις ε, σχέσεις με την Ανατολική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στιούαρτ. Και τώρα ερχόμαστε στον κύριο Λουμπασέγκο, ο οποίος είναι ε, ε, ερευνητής και blogger και έχει κάνει έρευνα για το θέμα της σύνδεσης στο διαδίκτυο και τη χρήση του διαδικτύου και των νέων μέσων στη μετασοβιετική ε, εποχή και στις μετασοβιετικές χώρες. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα ευκαιρία που μου δίδεται να συμμετέχω στην παρούσα ακρόαση και να σας παρουσιάσω μερικές ιδέες μου. Έχω κάνει κάποια έρευνα, γενικά βέβαια, ε, αλλά ιδιαίτερα και πρόσφατα στην επιρροή των νέων τεχνολογιών ε, στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες στις χώρες αυτές. Γι' αυτό θα σας μιλήσω και σήμερα. Έχω και κάποιες διαφάνειες ε, ετοιμάσει. Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το εξής ερώτημα. Γιατί το θέμα των νέων μέσων και η επιρροή τους ε, στην πολιτική ζωή των χωρών αυτών είναι το σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι το διαδίκτυο μπαίνει στις χώρες αυτές τις μετασοβιετικές πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία ε, για τις χώρες εταιρικής σχέσης και τη χρήση αυτή τη στιγμή. Ε, δεν υπάρχει κανένα τομέα της καθημερινότητας που να ξεφεύγει από τα like, τα tweets, τα σχόλια, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης κτλ. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό λοιπόν στι χώρε της Ανατολικής Κατά την άποψή μου οι πολιτικέ τη Ένωση προς τις χώρες αυτές ε, κυρίως στρέφονται προ τι ελίτ τη χώρα, ε, της εκάστοτε Υπάρχει κάποιο έλλειμμα σε σχέση με την άμεση επαφή, με την ίδια την κοινωνία, με τους πολίτες των κρατών. Ε, και η νέα τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει μια ευκαιρία να έρθουμε ε, πιο κοντά και να αντίνουμε την επικοινωνία μας με τις κοινωνίες αυτές και να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία και το κυβερνητικό επίπεδο, όπως ανέφερε η κυρία Στιούαρτ. Πώς επηρεάζουν λοιπόν τα νέα κοινωνικά μέσα αυτή την πραγματικότητα. Το διαδίκτυο δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι μόνο αισιόδοξο και θετικό. Από τη μια υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη πίεση για διαφάνεια, από την άλλη όμως είναι πιο δύσκολο για να μην πω αδύνατο να ελέγχουν οι κυβερνήσεις την κυκλοφορία των πληροφοριών. Και το διαδίκτυο στην μετασοβιετική εποχή και στο χώρο αυτό είναι ένα μέσο για τις κοινωνίες που έχουν ελεγχόμενο τύπο ή ε, μερικώς ελεύθερο για να έρθουν σε επαφή με κάποια ζητήματα που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να τους κρύβουν. Και επίσης ακούγονται και οι φωνές της αντιπολίτευσης και των πολιτικών που αποκλείονται από τα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης ή δεν έχουν καμία φωνή στον τύπο. Ξεκίνησαν κάποια αυθόρμητα κινήματα, είναι πολλά τα ε, παραδείγματα, δεν θα τα αναφέρω. Γνωρίζουμε επίσης ε, κάλλιστα ότι η τεχνολογία έχει και τη σκοτεινή της πλευρά και όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να ελέγχουν ε, αυτό το φαινόμενο που έχει λάβει διαστάσεις σαν ε, προηγουμένου. Δεν είναι άσπρο μαύρο η επιρροή της νέας τεχνολογίας. Υπάρχουν και κάποιες ε, σκοτεινές πλευρές που είναι κατακαιρματισμός της κοινή γνώμης, δεν υπάρχει κοινή πληροφόρηση σε μια ομοιόμορφη δηλαδή σε μια κοινωνία και υπάρχει και ένας ακτιβισμός Το βλέπετε στη διαφάνεια που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Ήταν το ε, ίντερνετ στην Ουκρανία αυτό πριν από λίγους μήνες. Κάτι άλλο σημαντικό Βεβαίως τα διαδικτυακά μέσα ε, είναι μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης από πλευράς κοινωνιολογικής και συχνά είναι και διασυνοριακά. Υπό την έννοια αυτή δίδεται η ευκαιρία να ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων ε, κοινωνιών στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Αλλά αυτό το καρπούται κυρίως η Ρωσία και το πρόγραμμα της για τα νέα μέσα. Κοιτάξτε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια πώς έχει η κατάσταση. Οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας ε, από το διαδίκτυο είναι μάλλον στη σφαίρα της ευρύτερης ρωσικής επιρροής και του ρωσικού κομματιού της φέτας στο διαδίκτυο. Επίσης δεν έχουν ξεκινήσει ε, νέα διασυνοριακά κινήματα, πλατφόρμες ε, νέων μέσων ε, στις χώρες αυτές που να είναι διασυνοριακές. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν επιμέρους στο εσωτερικό της κάθε χώρας και της κάθε κοινωνίας αλλά δεν έχουν ένα ευρύ αντίκτυπο στις γειτονικές χώρες. Άλλα σημαντικά ζητήματα είναι ε, τα εξής. Ενώ οι περισσότεροι πολίτες των χωρών αυτών θεωρούν ότι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και χωρίς λογοκρισία, χωρίς καταστολή. Ε, βλέπουμε πώς έχει η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία ε, του διαδικτύου. Δυστυχώς για τη Μολδαβία δεν έχουμε στοιχεία ούτε για την Αρμενία. Είναι λίγο ατελής αυτή η διαφάνεια. Προς το παρόν υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου χάσματος, μιας νέας διαχωριστικής γραμμής ε, σε αυτές τις χώρες ως προς τον κυβέρνο χώρο. Για μένα το πιο ανησυχητικό εμφανίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους στο Ντουμπάι σε μια παγκόσμια διάσκεψη τηλεπικοινωνιών ε, που ήταν ε, διαπραγμάτευση και υπογραφή νέων συμφωνιών και η διαχωριστική γραμμή ακριβώς διαπερνά τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, κυρίως Ουκρανία και Αζερβαϊτζάν. Φάνηκε ότι ήταν οι μόνες χώρες που υπέγραψαν αυτή τη νέα συμφωνία και τον κανονισμό. Ενώ η Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία ακόμα και Λευκορωσία ε, έμειναν εκτός την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό βέβαια δεν συνιστά ε, σε καμία περίπτωση απόδειξη για το προς τα που πηγαίνουν αυτές οι χώρες, αλλά μπορεί να εντοπίζει ένα πρόβλημα ε, στη σύγκληση τους ε, με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. οι οι χώρες που συντάσσονται με τη Ρωσία δηλαδή σε αυτό το τομέα δεν υπάρχει σύγκληση για ε, την κοινωνία της πληροφορίας διεθνώς και ε, σε σχέση με την Ανατολική γειτονία. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση διαφόρων κανονιστικών καθεστώτων και πλαισίων στις χώρες της Ανατολικής γειτονίας, να μην υπάρχει ομοιομορφία δηλαδή, ε, ούτε είναι δεδομένη η ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων χωρών ω προ το διαδίκτυο. Μερικέ προτάσει και ιδέε για το τι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα όφιλε να ε, πράξει ε, σχετικά. Πρώτον, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα ε, να μπει το θέμα της κοινωνίας της πληροφορίας ως μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ατζέντα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει και τα ίδια τα κράτη-μέλη και τους ανατολικούς γείτονες να ανταλλάσσουν πληροφορίες ε, ως προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που είναι ίσως ε, ένα από τα ε, πιο χρήσιμα εργαλεία για να επέλθει διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Επίσης και η διπλωματία μπορεί να ενισχυθεί από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνία με το κοινό. Θα πρέπει να ε, ε, υπάρξουν επενδύσεις ε, στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στις μετασοβιετικές χώρες για να έχουμε στοιχεία αξιόπιστα και ασφαλή Επίσης θα πρέπει να υποστηριχθούν κάποια έργα διασυνοριακής επικοινωνίας. Βλέπετε εδώ ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, μια πλατφόρμα νέων μέσων που δημιούργησαν Πολωνοί ε, φοιτητές. East Book EU ονομάζεται. Σε τέσσερις γλώσσες ήδη κυκλοφορεί και εκδίδεται αυτή η προσπάθεια. Υπάρχουν ε, και άλλα τέτοια παραδείγματα που αξίζουν και την προσοχή μας και την υποστήριξή μας. Και μακροπρόθεσμα θα άξιζε να σκεφτούμε μια προσέγγιση συνολική, ε, συνεκτική και ε, μακροχρόνια, αλλά βέβαια δεν είναι του παρόντος, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει ευρύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ συζητήσεις σας, για τις διαβουλεύσεις σας. Παρακαλώ τώρα τους συναδέλφους που έχουν στήσει το λόγο. Έχουμε κι άλλους. Θα πρέπει να τα πούμε πολύ γρήγορα γιατί μας μένουν μόνο 15 λεπτά. Κρόνμπεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η... Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις για την κυρία Στιούαρτ. Μιλήσατε πολύ για την κοινωνία των πολιτών και χαίρομαι που αυτό μπορεί να έχει και, το, και τον απόϊχό του ε, στην κοινωνία των πολιτών, αν και κάποιοι είπαν ότι δεν υπάρχει επαρκής επαφή. Ε, για την ασφάλεια όμως, τι έχετε να πείτε. Πώς βλέπει ο κόσμος την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιο βαθμό αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ε, θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βλέπουν σαν έναν εταίρο, τη βλέπουν σαν έναν εχθρό. Τι είδου ε, αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό δηλαδή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους για τις ε, τοποθετήσεις τους και θα ήθελα να ρωτήσω εάν παραλπίδα αναλάμβαναν καθήκοντα Πρωθυπουργού στο Βίλνιους. Λέτε ότι αυτή η εταιρική σχέση δεν δίνει τις ίδιες προοπτικές με αυτές που είχαν τα κράτη που έχουν εντωμεταξύ ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα έλεγαν λοιπόν όλοι αυτοί ε, οι κύριοι και οι κυρίες για να στηρίξουν την ε, η δυναμική των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών αυτών που βρίσκονται τόσο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται ε, υπό την επίδραση, την εξάρτηση από ένα τόσο μεγάλο εταίρο τη Ρωσία και πώς βλέπουν την εξέλιξη του πολυμερούς διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εταίρων προς τα Ανατολικά. Θεωρείται ότι οι πόροι οι οποίοι έχουν προβλεφθεί για το προσοχές πολιετές πλαίσιο της, ε, για την Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι επαρκής μπορούν να συντηρήσουν την δυναμική των χωρών αυτών και μια προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυρίλοφ, εντυπωσιάστηκα από την αναφορά στο ότι η πολιτική της αρεσιμότητας της επιβολής προϋποθέσεων για τις χώρες αυτές είναι όχι τόσο επιτυχής και ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και οι προϋποθέσεις. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κύριο που το ανέφερε να το επαναλάβει και να το αναλύσει. Και θα τον ρωτήσω εάν θεωρεί ότι θα πρέπει να ε, διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση μας προς τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να έχουμε αιρεσιμότητα ε, κατά περίπτωση. Γιατί υπάρχουν βέβαια διαφορές μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν χώρες στις οποίες μπορούμε να ζητήσουμε πιο φιλόδοξους όρους, άλλες με τις οποίες θα πρέπει να δείξουμε περισσότερη υπομονή. Και παρακαλώ τον ε, λόγο κύριο να αναλύσει τις θέσεις του. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Κύριο Στάνοκ, ε, εγώ θα ήθελα τις επόψεις των ε, ομιλητών ως προς ε, τις ως προς τη στάση των Ρώσων, της Ρωσίας και τον εκφοβισμό που επιβάλλει σε χώρες όπως ε, η Αρμενία, η Γεωργία και άλλες χώρες που θέλουν να προχωρήσουν με τις ε, συμφωνίες του Βίλνιους. Θεωρούν λοιπόν ότι η Ρωσία έχει καταστήσει στρατηγικό της στόχο να τις διατηρήσει ως δορυφόρους τους σε μια κατεύθυνση μάλλον πρώην Σοβιετικών κρατών ή θα τους επιτρέψει να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί αντιμέτωπη στη Ρωσία. Μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Μπορεί να δώσει περισσότερες, να κάνει πιο γενναιότερες προσφορές. Ή εάν η Ρωσία, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, απαγορεύσει την κυκλοφορία προϊόντων των κρατών αυτών. Την προηγούμενη εβδομάδα απαγόρευσε την κυκλοφορία ε, ίνου από τη Μολδαβία. Μπορεί και η, Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει ε, την κατανάλωση βότκας από τη Ρωσία Φερρυπίν σε αντίπεινα. Μπορούμε να έχουμε κάποια τέτοια μέτρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βουλιάνος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στην εξωτερική πολιτική και από την έκθεση αυτή βλέπω δύο, τύπων, δύο τύπους ε, γειτόνων να διακρίνονται. Εκείνους που για το ορατό μέλλον, ίσως και πιο μόνιμα θα είναι απλώς γείτονες, θα παραμένουν απλώς γείτονες, αλλά θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλοί γείτονες, να μην έχουμε προβλήματα μαζί τους. Και εκείνους οι οποίοι έχουν πιο προβεβλημένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, στους οποίους θα πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια, αλλά διαφοροποιημένοι. Τι πιστεύετε λοιπόν εσείς, οι χώρες της ανατολικής ε, γειτονίας σε ποια κατηγορία ανήκουν ή, να το πω αλλιώς, ανήκουν όλες στην ίδια κατηγορία ή μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Φυσικά το οικονομικό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν αποτελεί τον κύριο παράγοντα παροχής βοηθείας προς τους γείτονες ώστε να έρθουν πιο κοντά σε εμά. Θα μπορούσαμε να τους ενθαρρύνουμε φερρυπίν με ε, την ε, υποδειγματική μας τάση, με την καλή πρόθεση και διάθεση που θα δείχναμε, με την υποστήριξη έναντι των πιέσεων οικονομικών, διπλωματικών και άλλων της Ρωσίας. Και σε μια ιδιαίτερη κατάσταση δεν νομίζετε ότι το πιο σοφό στην προκείμενη περίπτωση θα ήταν να ανοίξουμε πιο ευρύ διάλογο με τη Ρωσία και να πείσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι είναι στο δικό, για το δικό της συμφέρον, είναι προς το συμφέρον της να αφήσει χώρες ελεύθερες να εκφράζουν ελεύθερη βούληση και να επικοινωνούν ή να αναπτύσσουν σχέσεις όπως θεωρούν σκοπιμότερο, με οιονδήποτε θεωρούν σκοπιμότερο. Η αφύπνιση των κρατών αυτών και υποστήριξη της αφύπνισης των κρατών αυτών. Ο στόχος της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός πιστεύω, άλλωστε και οι ομιλητές μας επισήμαναν ότι υπάρχουν τα σχετικά εργαλεία. Και ρωτώ εάν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε κάτι επιπλέον, βράχη πρόθεσμα, ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των κρατών αυτών, η αυτοσυνείδηση ότι είναι όντως ευρωπαϊκά κράτη. Благодаря. Χωρίς μικρόφωνο, μίλητης Η κυρία Λιουμτσέφα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ήταν ευρύτατη η βάση συζήτηση προσφέρουν οι αναλύσεις τους. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή μας μέσα αυτό το μήνα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο για τη συζήτηση ε, για την Ανατολική Γειτονία, όπως έχει ήδη πράξει. Άλλωστε πολλά έχουν υποθεί και πολλά επαναλαμβάνονται στις συζητήσεις μας. Πρέπει να συνεχίσουν όμως συζήτησεις για την Ανατολική κοινωνία. Εγώ βλέπω σήμερα ότι η κατάσταση φαίνεται να μας οδηγεί στην αναζήτηση πιο συγκεκριμένων ε, στήριγμάτων όπως η Ουκρανία. Γι' αυτό τον κύριο Αντάμσκι θα ήθελα να ρωτήσω ε, ω ειδικό τι είδους ε, μέτρα, τι είδους βήματα θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό ποιες συνθήκες ώστε να προβάλλει την ε, συμφωνία, να προωθήσει τη συμφωνία για, τη σύνδεση με την Ουκρανία. Για το Βίλνιους τι μπορούμε να περιμένουμε και έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η κοινωνία των πολιτών εξελίσσεται και στη δική μου την πατρίδα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και βλέπω πως η κοινωνία των πολιτών και στα κράτη της Ανατολικής ε, Γειτονίας χρειάζεται πολύ προσεκτική θεώρηση και ανάλυση. Πώς βλέπετε λοιπόν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είναι ουδέτερες και ακομάτιστες και μπορούν να συνδεθούν σε ε, πολιτικά εγχειρήματα και σχέδια. Βλέπετε αυτό να αποτελεί μια εξέλιξη ε, προ όφελο των πολιτών και όχι μια εξέλιξη που όπως εξυπηρετεί κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές ελίτ. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ έχω να κάνω ορισμένες ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις στα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Η πιο σημαντική καταρχήν ε, νομίζω είναι φανερό ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έναν τομέα διείσδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές. Το είδαμε και σήμερα. Λες και οι χώρες αυτές και οι λαοί αυτοί δεν έχουν να προσφέρουν κάτι ε, αναπαράγεται το υπερρεαλιστικό να πάμε του εκπολιτίσουμε με έναν τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας ε, εμεί είμαστε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σχέσεις ισότιμες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπιέται με τη Ρωσία για ζώνες επιρροή στις χώρες αυτές. Η ερώτηση μου είναι εξής. Από τα στοιχεία που μας έδωσε ο κύριος για τη διάδοση του διαδικτύου του ίντερνετ φάνηκε ότι η επιρροή της Ρωσίας είναι να πούμε πιο μεγάλη από ό,τι αυτή των Δυτικών. Αυτό βέβαια έχει ιστορικούς λόγους και άλλους λόγους. Και παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι σχετικά ελεύθερο, βλέπετε ότι οι προτιμήσεις του κόσμου είναι προς Ανατολάς. Δεν έχω καμία προτίμηση για τη Ρώσικη Ομοσπονδία. Κάθε άλλο μάλιστα γιατί και εκεί αναδεικνύεται μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη. Όμως, το ερώτημα που υπάρχει είναι έχει επίγνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλουν οι λαοί αυτών των χωρών, τι ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διαμορφώσει όσο μπορεί περισσότερο ισότιμες σχέσεις ή απλώς πάει με μια δική της πολιτική, κάνει την πολιτική άρσης της ε, ε, θεώρησης διαβατηρίων για να προωθηθεί βέβαια η κινητικότητα αλλά και το brain drain για το οποίο δεν έγινε συζήτηση και από εκεί και πέρα, εν και οι χώρε αυτέ α μείνουν σε συνθήκε οικονομική κρίση σαν και αυτέ και χειρότερε που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Ε, very brief comment. Εντάχει, διότι πρόκειται για μία συζήτηση στο Δινεκές για την πολιτική γειτονία, ιδιαίτερα στο Στρασβούργο. Η συζήτησή μας σήμερα αφορά μια πολιτική γειτονίας που έχει λήξει, γιατί πολλοί δεν έχουν αποφασίσει ε, σε σχέση με την προσχώρηση στην Τελωνιακή Ένωση και αυτό που έχει σημασία είναι να ορίσουμε μια νέα πολιτική γειτονίας σε αυτούς που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και ορισμένες ε, χώρες προσχώρησαν στην Τελωνιακή Ένωση πρωταρχικά, διότι η Ρωσία δεν ασχολείται μόνο με την Τελωνιακή Ένωση, ε, προσβλέπει ίσως ένα πρότυπο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε χώρες όπως ε, την Αρμενία. Διότι η περίπτωση αυτή καταδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με μία νέα ε, πραγματικότητα σε σχέση με την ε, παλαιά μας φιλική πολιτική, η οποία βαίνει στο τέλος της. Ε, πολλές φορές υπάρχουν θετικές εκβάσεις, άλλες λιγότερο. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Έλληνα συνάδελφο, ο ναι. οποίος έλαβε το λόγο. Δεν δέχομαι αυτή τη γλώσσα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε αντιπαλότητα με τη Ρωσία ή σε αντίθεση. Η Ρωσία είναι εκείνη η οποία ε, διαπραγματεύτηκε με την ελεύθερη Ευρώπη, με τους ελεύθερους ανθρώπους. Αν δείτε το καθεστώς ε, θεωρήσεων και πώς ορίζεται, μπορείτε να δείτε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προσφέρουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο ε, αυτό το πλαίσιο δεν ήταν λειτουργικό στην Πολωνία την περίοδο του ε, κομμουνισμού. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε στην Ελλάδα, αλλά δεν δέχομαι τη συλλογιστική που προέβαλε ο Έλληνας συνάδελφος πρόσφατα ότι κατανοώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν μία κοινή βάση και θα ήθελα να δώσω ε, μία απαρχή απάντησης στις ερωτήσεις αυτές. Όπως είπα στην παρουσίασή μου εξ αρχής, η ανατολική ε, εταιρική σχέση είναι ένα ελιτίστικο πρόγραμμα, διότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ε, κοινωνιών πάντα. Γι' αυτό όταν αυτές οι χώρες ε, λάβουν τις αποφάσεις τους προς τα που θα κινηθούν, θα είναι δική τους η απόφαση που θα βασίζεται σε αυτές σε αυτές τις ε, κοινωνίες. Δημοκρατικά ή μη δημοκρατικά καθεστώτα έχουν αυτές τις εταιρικές σχέσεις και αυτές οι ελίτ πρέπει να λάβουν υπόψη την ε, κοινή γνώμη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει σε αυτές τις σφαίρες ε, επιρροής θα πρέπει να συνεργαστεί με την κοινή γνώμη. Τώρα ποια είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις χώρες Κανείς ε, εξ αρχής δεν θεωρεί εχθρό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λάβετε υπόψη την ε, Ουκρανία που είναι και η πιο κοντινή για μένα, οι έρευνες έχουν ε, δείξει ότι η κοινωνία υποστηρίζει την στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η κοινωνία δεν ξέρει έμπρακτα τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ολοκλήρωση Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το επεξηγήσουμε. Καταρχήν στην κοινή γνώμη, στους αρχηγούς και να διαδώσουμε αυτή τη μορφή κατανόησης. Αυτή είναι η απάντηση στις ερωτήσεις αυτού του τύπου. Ας προσπαθήσουμε οι κοινωνίες να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα και ας αποφασίσουν μόνες τους. Ε, έλλειψη συμφωνιών δεν σημαίνει και έλλειψη συνεργασίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την διαδικασία. Δηλαδή προσβλέπουμε σε συμφωνίες μέσα στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πιο παραγωγικά με αυτές τις ε, χώρες. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Στιούαρτ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ. Τώρα, ε, δεν ε, θα μιλήσω για τη βότκα και ε, άλλα ποτά, για το κατά πόσο πρέπει να εισάγεται ή όχι. έχω μια ερώτηση στον κύριο Αντάμσκι και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Μιλήσατε για έλλειμμα επικοινωνίας στην Ουκρανία. Έχετε διαπιστώσει. Αυτό ισχύει και για τη Συμφωνία Σύνδεσης, να γνωρίζει ο κόσμος και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει αυτή την άγνοια. Και μια άλλη ερώτηση μιλήσατε για ρωσική πίεση. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι και μια ε, αποτροπή από το να ε, προχωρήσουν στην Ευρασιατική Ένωση. Τι ε, μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το αντικρούσει αυτό. Και έχω και μια ερώτηση προς την κυρία Στιούαρτ. Αυτό το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών τι επιπτώσεις έχει στις χώρες ανατολικής γειτονίας. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα κατά πόσο συμμετέχει η Λευκορωσία. Μια χώρα με την οποία έχουμε πάρα πολύ τεταμένες ε, σχέσεις. Και είναι κάπως ε, ικανοποιητική ακόμα η συνεργασία με το Φόρουμ Πολιτών. Εσείς πώς εκτιμάτε τις επιπτώσεις και τις επιρροές στις διάφορες χώρες, κυρία Στιόρτ. Ευχαριστώ. Καταρχήν το θέμα που εφήγει ε, πριν απαντήθηκε από τον κύριο Λουκασένκο. Δηλαδή κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται συνεργάτης ή εχθρός. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ε, συνεργατικός εταίρος ε, ένας από τους πολλούς εταίρους, διότι οι χώρες αυτές επιφυλάσσονται και πριν προβούν σε αυτή την επιλογή ε, θέλουν να έχουν συνεργατικά σχήματα με όλες τις χώρες και με τη Ρωσία. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι Ευημερία, το οποίο δεν ισχύει με την ε, ναι. τρέχουσα, υπό την τρέχουσα ε, κρίση, αλλά η ευημερία σημαίνει και προστασία πολλών δικαιωμάτων. Σε σχέση με τη συστάδα των ερωτήσεων για το ρόλο της Ρωσίας και την αιρεσιμότητα, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε δύο τομείς και θα πρέπει να ξαναδούμε την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας. Όχι μόνο εξαιτίας της τρέχουσας ε, δραστηριότητας της Ρωσίας έναντι των γειτόνων, αλλά και λόγω των ε, εσωτερικών εξελίξεων της Ρωσίας αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προωθηθεί η ανατολική συνεργατική σχέση, η οποία δεν είναι ένα γεωπολιτικό μέσο και στόχο έχει να υπηρετήσει όλες τις χώρες. Νομίζω ότι η αιρεσιμότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συνεπή στην προσέγγιση της προς τις χώρες της ε, ανατολικής ε, αυτής της ε, συνεργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Σε σχέση με την επερχόμενη απόφαση στο Βίλνιους για την συνεργασία με την Ουκρανία και τη Συμφωνία Σύνδεσης, η Ρωσία μερικές φορές ε, απειλή. Η Ρωσία θέλει στρατηγικά να κρατήσει αυτές τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πιστεύω ότι η Ρωσία πια δεν έχει αυτό το στόχο, τουλάχιστον φαίνεται από τις ε, πρόσφατες δράσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να υπάρξουν ε, αντικρούσεις και αντισταθμίσεις του είδους ότι δεν θα πρέπει να εισάγουμε ρωσική βότκα υπομορφή αντιπίνων. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τις διάφορες συμφωνίες και σχήματα όπου συμμετέχει η Ρωσία. Αυτό αφορά και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Άρα, ε, ως προς την Ουκρανία, η απόφαση περί υπογραφής ε, αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πέρσι το Δεκέμβριο και δεν σχετίζεται με γεωπολιτικούς ε, συσχετισμούς. Ως προς την ερώτησή σας για τις επιπτώσεις των ε, φόρα της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους, νομίζω ότι η επιρροή είναι περιορισμένη και υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα φόρματ που είναι ελιτίστικα μέσα στα πλαίσια των ΜΚΟ, όπως είπε και ο κύριος ε, Λουκασένκο, υπάρχουν, ε, υπάρχει αυτή η ελιτίστικη προσέγγιση και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περισσότερο για να υπάρξει ένα σύνδεσμος μεταξύ αυτών των φόρων και των κοινωνιών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, σε σχέση με τη, τα κίνητρα και την ε, ανάπτυξη της οικονομίας σημαίνει ε, καταρχήν ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου δεν είχαν, στήχη, δεν είχαν τύχη σωστής ερμηνείας, κάτι το οποίο όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε προς, προς την Ουκρανία, με, με την Αρμενία με συγχωρείτε, ε, τέθη ένα ξεχωριστό ερώτημα. Η Αρμενία θα προσχωρήσει στην Τελωνιακή Ένωση κατά πάσα πιθανότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και της ε, καλύτερης, ε, της πιο προωθημένης εμπορικής συνεργασίας συν ε, την κινητικότητα. Η ρυθμιστική προσέγγιση, η οποία είναι συμπεριληπτική, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα θέσει στην άκρη ορισμένα ζητήματα, οι πτυχές αυτών. Αυτό που έχει σημασία είναι η συλλογιστική των γειτόνων χωρών και πολλές φορές η προσέγγιση είναι διαφοροποιημένη. Εδώ αναφέρομαι στο βάρος της ιστορίας Ορισμένες χώρες δεν μπορούν να προσεγγίσουν τις πλέον αναπτυγμένες χώρες και αυτό εξαρτάται από κάθε χώρα ξεχωριστά. Έχει σημασία λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι η αιρεσιμότητα που θα χρησιμοποιήσουμε επικεντρώνεται σε επιμέρους ζητήματα. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ασχολείται επί δεκαετίες με αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να μεταχειριστούμε όλους τους πελάτες ε, κατά τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να ορίσουμε σε κάθε χώρα ποιος είναι ο απαράβατος όρος για την πρόοδο. Ο εκφοβισμός της ε, Ρωσίας θα είναι αντιπαραγωγικός, αυτή η τακτική δηλαδή που ακολουθεί η Ρωσία. Στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγήσει σε μία καθαρά εκπτωτική σχέση. Πολλές φορές βεβαίως η Ρωσία προβάλλει αντιπαραγωγική, μία αντιπαραγωγική τακτική την οποία στη συνέχεια εγκαταλείπει. προβάλλοντας ε, διάφορες δικαιολογίες. Τώρα η σχέση μεταξύ Τελωνιακής Ένωσης και πιο στενών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκη. Ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους πάγιους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και να μην εφεύρουμε κάτι το εξολοκλήρου καινούριο. Η κυρία Στιούαρτ μίλησε και για το ρόλο του ΠΟΕ σε σχέση με τον εκφοβισμό από πλευράς Ρωσίας, αυτή την τρομοκρατία από πλευράς Ρωσίας. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να, ε, να υπάρξει ε, μία ε, πολύ καλή ατμόσφαιρα με τις γείτονες χώρες Ανατολών, αλλά να επέλθει μία πραγματική αλλαγή σε αυτές τις χώρες, να την επιβάλλουμε να ισχύσει μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Βεβαίως χρειάζονται περισσότερα κονδύλια, αλλά αυτό ε, πολλές φορές δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το DCFTA που είναι ένα, το πραγματικό μέσο, ουσιαστικό μέσο και η απαλληφή των θεωρήσεων η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι τα μόνα μέσα τα οποία θα οδηγήσουν σε πραγματικές αλλαγές της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αυτή είναι και η σύμβουλή μας. Τώρα, τι θέλει η Ουκρανία, τι θέλει η κοινωνία των πολιτών σε σχέση με τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι 45-50% της κοινή γνώμης της Ουκρανίας επιθυμεί μία συμφωνία σύνδεσης και ένα 35% επιθυμεί την Τελωνιακή Ένωση με τη Ρωσία. Όμως οι νέοι θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και η γυρεότερη γενεά είναι υπέρ της Τελωνιακής Ένωσης με τη Ρωσία μόνο, όμως το 20% ε, ε, ταυτίζεται με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μία δύναμη η οποία αποδομείται. Και αυτό αποτελεί πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πώς θα αντιδράσει και τι μέτρα θα λάβει, τα οποία δεν είναι πάντα φιλικά και ευπρόσδεκτα. Δεν βλέπω άλλη επιλογή παρά τον διάλογο με αυτή τη ρωσική ελίτ, το οποίο δεν είναι κάτι το μοναδικό. Ε, όχι όμως αντιπερισπασμούς ε, του τύπου απαγόρευσης εισαγωγών ε, βότκας από τη Ρωσία. Κάτι το οποίο δεν θα γινόταν κατανοητό από την κοινωνία της Ρωσίας επίσης. Θα πρέπει να θεωρήσουμε τη Ρωσία συμβαλόμενο μέρος ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων μέσα στα πλαίσια του, της τρέχου υπάρχουσες ε, νομική σχέσης που μας διέπει. Και ακόμα να απαντήσω σε μια ερώτηση στα γερμανικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τα ζητήματα της έλλειψης ενημέρωσης ως προς τα ελλείμματα. Νομίζω καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη πολιτική για τις θεωρήσεις, πιο ευφυείς υπαλλήλου στα προξενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ενημερώσουμε, για, για να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα ενημέρωσης. Σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, να ενημερώσουμε περισσότερο. Η Κουρανία, παραδείγματι, έχει αυτή τη στιγμή πολλές διαφημίσεις που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία χώρα με μία μόνο γλώσσα, τα αγγλικά, με μία μόνο οργάνωση κεντρική. η οποία περιορίζεται μόνο στην προαγωγή των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων. Αυτή είναι η εικόνα που δίνεται από τις διαφημίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω του τύπου στην Ουκρανία μέσω του διαδικτύου. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η ενημέρωση για την Ουκρανία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία και βέβαια μια καλύτερη πολιτική και πιο ευφύης πολιτική για τις θεωρήσεις. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Όσο μπορείτε να έχουμε και το γραπτό κείμενο, θα ήταν χρήσιμο. και ίσως και μετά το Βίλνιους ήταν σκόπιμο να παραμείνουμε σε επαφή. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σας, για την ενημέρωση που μας προσφέρατε. Ο κύριος Αγκουράκης νομίζω στάει το λόγο για άλλη μια φορά. Ο κύριος Αγκουράκης στάει το λόγο για άλλη μια φορά νομίζω, όχι. Θέλω να πω στον κύριο Αγκουράκη εγώ ότι είμαστε ε, πάντοτε υπέρ των ίσων δικαιωμάτων και αυτό είναι και η διαφορά σε σχέση με την Ρωσία. Τις, αποτελε... τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνει όσο αφορά εμάς ε, ούτε η Ρωσία, ούτε η Μόσχα δηλαδή, ούτε οι Βρυξέλλες, αλλά η κάθε χώρα μόνη της, η Τυφλίδα και ούτω καθεξής, η κάθε κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν σε σχέση με τη θεώρηση ε, τη δική μας. Σας ευχαριστώ. hope you too. Hello, Mr. Brock. Hello, hello. Meine Damen und Herren, ich darf Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στη μέσα διάταξη. Από, μαζί με τους συναδέλφους ε, από τις αντιπροσωπείες ε, Αζερβαϊτζάν, Αρμενίας και Γεωργία είναι ένα σύνολο κρατών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές εξελίξεις αυτή η ομαδοποίηση. Λοιπόν, παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία. Tanya, could you please leave the room? Λοιπόν, παρακαλώ σταματήσουν οι ιδιωτικές συνομιλίες. I would like Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω ενώπιόν μας την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας, οι πρόσφατες εξέλιξεις στη Γεωργία ιδιαίτερα ε, ως προς τη δικαιοσύνη αλλά και ε, προετοιμάζοντας ε, τη διάσκεψη του βίλνιου είναι το θέμα μας. Καλωσορίζουμε την κυρία Τσούλου και Άννη. Η ανταλλαγή απόψεων είναι επίκαιρη και πρόσφορη εν ώψη και των προεδρικών σας εκλογών αλλά και τη διάσκεψης κορυφής του Βίλνιου. Και επίσης βλέπουμε και τη Ρωσία να ασκεί κάποια πίεση Και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο νομίζω κάναμε ένα αρκετά καλό ψήφισμα σχετικά. Η κυβέρνηση πλέον έχει συμπληρώσει ένα έτος ε, στην εξουσία. Έχει έρθει η ώρα ενός πρώτου απολογισμού. Ε, ήταν μεγάλη σας προτεραιότητα η ε, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και πρόσφατα ολοκληρώσετε την πρώτη φάση. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μοιραστείτε μαζί μας ε, τα αποτελέσματα αυτά, καθώς επίσης και τι απομένει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επιλεκτική ή την πολιτικά κινούμενη δικαιοσύνη. Ε, σε αρχές Ιανουαρίου ε, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Η Επιτροπή της Βενετίας έχει εκφράσει μεγάλες επιφυλάξεις για την ανάμειξη μη δικαστικών σωμάτων στη δικαιοσύνη, πράγμα που ε, θέτει ένα αμφιβόλο το σύνολο της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ιδιαίτερα... κάποιες καταγγελίες είναι πιο πρόσφατα να γίνουν στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Έχουν γίνει κάποιες υποκλοπές, κάποιες παράνομες ε, ε, μαγνητοφωνήσεις, ευρέθησαν πρόσφατα και κατεστράφησαν. υπάρχει και μια προσπάθεια για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Μπορείτε να μας ε, ενημερώσετε για το κλίμα γενικότερα στη Γεωργία και τι συμβαίνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μετά από μεγάλη πίεση της κυβέρνησης, λέει, ε, παρετήθηκαν κάποιοι δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια και τον επόμενο Μάιο θα γίνουν δημοτικές εκλογές για να αλλάξει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, ανησυχούμε για την κατάσταση ε, σε ε, ένα δήμο που έγιναν ταραχές και ε, υπήρξαν προβλήματα μετά από την απομάκρυνση ενός μιναρέ. Είπατε ότι θα ε, παρετηθείτε μετά τις προεδρικές εκλογές. Τι σημαίνει αυτό ε, για τη συνέχεια στην πολιτική της χώρας σας. Κυρίως θα ήθελα να μας δώσετε την ερμηνεία σας για την κατάσταση στη χώρα τι γίνεται με την Τελωνιακή Ένωση, δεν έχει ληφθεί απόφαση, αλλά θα μας ενδιαφέρε να μάθουμε τις απόψεις. Θα ήθελα να σας πω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να επιτύχει η Σύνοδος Κορυφής στο Βίλνιος και γι' αυτό ελπίζουμε να υπάρξει δυνατότητα να μονογραφηθεί αυτή η συμφωνία με τη χώρα σας. Νομίζω το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί. Ελπίζω να μας βοηθήσετε κι εσείς στη διαδικασία αυτή. Έχετε καλό το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, για μένα είναι τιμή να έρχομαι εδώ, ε, να απευθύνομαι στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να σας παρουσιάσω την κατάσταση της Γεωργίας ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία και τις φιλοδοξίες της, καθώς επίσης και εν ώψη ε, ε, τη Συνόδου Κορυφής του Βίλνιου στα θέματα της γειτονίας. Έχουμε προκλήσεις ε, και δοκιμασίες στη διαδικασία αυτή τώρα. Διαπιστώνουμε και εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι μας υποστηρίζετε και εσείς και ο πρόεδρός σας ε, πριν από μία εβδομάδα στο Βίλνιου στην άτυπη ε, συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης για τη Συρία. Όλοι οι δρόμοι προς την Ευρώπη περνούν από το Βίλνιους. Ωστόσο, η δική μου πρόθεση δεν είναι να κάνω άλλη μια πολιτική δήλωση, αλλά να σας πω ότι φέρνουμε επιτάπητος ε, στην ατζέντα και στα κοινά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ως υπουργό Δικαιοσύνης και μέλος της κυβέρνησης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το μέλλον της γεωργίας, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Βασικός μας στρατηγικός στόχος είναι και παραμένει ε, η ευρωπαϊκή πορεία. Να έχουμε μια θεσμική δημοκρατία, δηλαδή να δημιουργήσουμε ε, τις προϋποθέσεις για πολιτική σύνδεση και οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό να είναι τόσο στέρεο ώστε να μην μπορεί καμία κυβέρνηση να το αποδομήσει. Ο εξευρωπαϊσμός της χώρας να είναι μη αντιστρεπτός. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ε, υλοποιήσουμε τις ε, δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις μας, να ευθυγραμμιστούμε με ευρωπαϊκούς κανόνες και πολιτικές. Ε, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως ονομάζεται κανονιστική δύναμη. Στη Γεωργία ε, το αντίστοιχο είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται και η κυβέρνηση, καθώς επίσης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προσφέρει πολλές φόρμες για ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του κοινού σε αυτή τη διαδικασία. Δεν περιορίζουμε ε, κανέναν, είναι ευρία συμμετοχή σε δημόσιες συνεδριάσεις, ακόμα και άμεση επικοινωνία έχουμε με ε, το λαό για τη λήψη των αποφάσεων. Δεν υπάρχει ούτε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που να ε, μην υποβάλλεται, ε, μάλλον, που να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο χωρίς να έχει υπάρξει πρώτερη δημόσια διαβούλευση. Γενικώ ε, έχουμε ελευθερία στην ενημέρωση, δημόσια διαβούλευση εκ των προτέρων πριν κατατεθεί κάθε νομοσχέδιο, ε, και όλα αυτά στα πλαίσια της ε, ανοιχτής διακυβέρνησης της Γεωργίας. Όλο και περισσότερο πιστεύουμε ότι μπορεί να μονογραφηθεί στο Βίλνιους η Συμφωνία Σύνδεσης και να υπογραφεί πριν τα τέλη ε, της θητείας παρούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε αρχίσει ήδη να προσεγγίζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο με κάποιες νομοθετικές αλλαγές πολύ πριν ε, λάβουμε την ατζέντα για τη σύνδεση. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο που καταρτήσαμε πρόσφατα για τη χρηματοδότηση της νομοκρατίας. Έχει ήδη σταλεί στο Κοινοβούλιο. Αυτό τον καιρό συνεργαζόμαστε ε, και εργαζόμαστε για την ε, Συμφωνία Σύνδεσης για να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμόζεται σωστά αφενός και αφετέρου να είναι και ένα τμήμα του ε, σύνολου θεσμικού μας και συνταγματικού πλαισίου. Να υπάρχουν συνταγματικέ συνταγματικές εγγυήσεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας. Έχει επιτευχθεί πρόεδρος επίση και στην πρώτη φάση του προγράμματο δράση για την απελευθέρωση απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, όπου πρωτοστατεί το Υπουργείο μας μαζί με άλλα Υπουργεία. Για παράδειγμα, για τον νόμο κατά των διακρίσεων, που έχει ήδη καταρτιστεί το νομοσχέδιο και έχει σταλεί ε, για ε, διεθνή ε, έλεγχο, η καταπολέμηση ε, της διακίνησης ανθρώπων, της διαφθοράς, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση, είναι άλλα θέματα που μας απασχολούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι μέσα Οκτωβρίου να έρθει η αποστολή εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περάσουμε στη δεύτερη φάση. Ο νόμος κατά των διακρίσεων είναι πολύ καλό νομοσχέδιο που βασίζεται την ευρωπαϊκή εμπειρία και τις διεθνείς προδιαγραφές. Έτσι στο μέλλον δεν θα εμφανίζονται φαινόμενα και καταστάσεις σαν αυτές που περιγράψατε πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη Τσέλα. Ε, δημιουργείται ένα ισχυρό πλαίσιο ε, ισότητας, αντιμετώπιση των διακρίσεων, ε, συστηματοποιείται ε, η νομοθεσία που ήδη υπάρχει για τις διακρίσεις, τα πολέμησή τους. Ας πούμε, η αναπηρία είναι κάτι που δεν αναφέρεται στο νόμο. Η, η μητρότητα, η εγκυμοσύνη, ο ε, σεξουαλικός προσανατολισμός, η ιδιότητα του φίλου Έχουμε μια προοδευτική προσέγγιση για την ε, καταπολέμηση όλων των διακρίσεων και μάλιστα των πολλαπλών διακρίσεων και αυτό είναι κάτι το ε, πολύ σύγχρονο σε σχέση με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης οι διάφοροι ε, φορείς ε, διορίζονται ε, με κριτήρια μη πολιτικά και με συμμετοχή του Κοινοβουλίου και με εξαρτησία πάντα και νομική και οικονομική. Αυτός ο νόμος θα προκύψει μετά από την ευρεία διαβούλευση αφού θα έχουν εκφράσει τη γνώμη τους και εξακολουθούν να την εκφράζουν όλοι οι ενεχόμενοι και ενδιαφερόμενοι. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο διπλωματικό σώμα και στην κοινωνία των πολιτών στις διάφορες θρησκευτικέ ομολογίες καθώς επίσης και εθνικές μειονότητες των οποίων ζητήθηκε η γνώμη. Και στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υποβληθεί και σε Σουηδό εμπειρογνώμονα και τελικά θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Προεδρικές εκλογές. Ε, σε ένα συνταγματικό πλαίσιο έχουμε αλλαγή της εξουσίας και πέρσι τον ε, Οκτώβριο άλλαξε η κυβέρνηση. Οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές είναι πραγματικά δοκιμασία και λιδία λήθος για τη δημοκρατία στη Γεωργία. Για να γίνει με τρόπο ε, διαφανή και δίκαιο και ελεύθερο αναμέτρηση αυτή έχει ε, δημιουργηθεί αντίστοιχη επιτροπή με εντολή να ε, προλάβει ε, τις παρεμβάσεις με ειδικέ συστάσεις. Επίσης έχει ήδη ασκήσει τα καθηκοντά της, έχει κάνει συστάσεις σε όλους τους μεγάλους θεσμούς και τους μεγάλους ε, που είναι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Υπουργεία, Πολιτικά Κόμματα, Όργανα επιβολή τη τάξη, ε, Οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να παρακολουθεί την προεκλογική καθώς και την εκλογική διαδικασία και ε, θα προτείνει και θα λάβει τα αντίστοιχα μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων. Εγώ προεδρεύω σε αυτή την Επιτροπή και πολύ πρόσφατα μετέβη σε μία από τις περιφέρειες όπου υπήρξαν κάποιες μεταθέσεις προσωπικού ανησυχητικές. Εξέφρασε ανησυχίες κοινωνία των πολιτών. Χάρη στις δικές μας συστάσεις η κατάσταση σήμερα σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σταθερή και οι πάντες κατέλαβαν, ότι οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες. Πέρυσι η Γεωργία κατάφερε να μεταφέρει ε, την εξουσία από το ένα κοινοβούλιο στο επόμενο με ειρηνικό τρόπο και τώρα αυτό που αναμένεται να αλλάξει μέσα από εκλογές είναι ο πρόεδρος χωρίς καμία βία. Το σημερινό περιβάλλον, το προεκλογικό, είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που γνωρίσαμε ε, στο παρελθόν. Και θυμάμαι εγώ γιατί ήμουν υποψήφια ε, πέρυσι, τον Οκτώβριο, τι γινόταν η δικαιοσύνη είναι το σημαντικότερο και το πρώτο θέμα και προτεραιότητα για τις μεταρρυθμίσεις και για την υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2017. Επικεντρωνόμαστε στις θεσμικές εγγυήσεις για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των μεμονωμένων δικαστών με βάση την αρχή more for more, περισσότερα, με αντάλλαγμα περισσότερα και θα πρέπει τακτικοί δικαστές να εργάζονται σε ένα σωστό πλαίσιο, καθώς επίσης και το Ανώτατο Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης. Είναι ένα νέο συσταθένο όργανο αυτό, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και είναι ακριβώς η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και των μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε πριν από μία εβδομάδα για τον τρόπο διορισμού, προαγωγής και ε, ανάθεσης διαφόρων υποθέσεων σε μεμονωμένους δικαστές. Ε, ο κώδικας ποινική ε, δικονομίας και τα διοικητικά ζητήματα θα αναθεωρηθούν επίσης μέχρι τα τέλη του έτους. Τα δικαιώματα των θυμάτων θα μισθούν με την ευρωπαϊκή ε, πραγματικότητα και επίσης η δικαιοσύνη που αφορά τους ανηλίκους είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δημιουργηθούν ξεχωριστά δικαστήρια ανηλίκων. Επίσης η εισαγγελία ε, χρειάζεται μεταρρύθμιση για να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος και η ανεξαρτησία της εισαγγελίας για να μπορεί να λειτουργεί με τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό όσο και επαγγελματικό. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα. Όλες οι εξουσίες που ήταν στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης έχουν μεταφερθεί τώρα στο Γενικό Εισαγγελέα. Εγώ δίωξης δηλαδή. Οι ε, βασικοί εισαγγελεί πλέον είναι ανεξάρτητη από την πολιτική, από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και από οποιαδήποτε πολιτική επιρροή. Ε, ένα άλλο νομοθετικό πακέτο αφορά τη σταδιακή διεύρυνση ε, της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων για κάποιο είδους κακουργήματα και τη συμμετοχή των πολιτών στη διοικητική μηχανή, έτσι ώστε να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα. Η μεταρρύθμιση μας βασίζεται σε σωστή χρηματοδότηση, σε σωστά προγράμματα, ε, δράσεις με ε, κατάλληλο συνδυασμό με στόχους χρονικούς δείκτες ε, και παρακολούθηση. Αυτά τα προγράμματα δράσης αυτό το καιρό ανανεώνονται για να δώσουν μια νέα εικόνα και ένα νέο όραμα για τη δικαιοσύνη μας στο επόμενο διάστημα. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να πω το εξής και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω λεγόμενα φαινόμενα κακοδικίας. Διάφορες μη νομικοί εμπειρογνώμονες, ε, γεωργιανοί καθώς και αλλοδαποί καταγγέλουν τέτοια θέματα και πήραμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βενετίας ε, και λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά ε, τα θέματα και όλες τις συστάσεις που περιέχονται. Ο νόμος αυτός δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα δικαιοσύνης που οικοδομείται αυτή τη στιγμή στη Γεωργία. Αυτός ο νόμος σημαίνει ότι χιλιάδες Γεωργιανοί θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ε, αίτηση σε μια επιτροπή ε, που θα είναι εκλεγμένα τα μέλη της από την κοινωνία των πολιτών με ε, προφανώς ε, πραγματογνωμοσύνη και βοήθεια νομική και από το Κοινοβούλιο. Και αν θέλει, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και ο δικαστής θα έχει τον τελικό λόγο για μεμονωμένες ποινικέ υποθέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να απευθύνονται στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου γιατί αυτές οι υποθέσεις έχουν ξεφύγει από το εξάμεινο χρονικό περιθώριο. Ο Πρωθυπουργό και η παρέτησή του μάλλον ε, μας ήρθε ε, ως μια πολύ κακή είδηση ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ζήτησε την υποστήριξη όλων των μελών και είμαστε πρόθυμοι να τον βοηθήσουμε να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις ε, και τις πολιτικές και τις δικαστικές, αφού το ανέλαβε και μετά τις προεδρικές εκλογές ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό με το πιο διαφανή τρόπο. Να μπορέσει να αποχωρήσει ο Πρωθυπουργό και να αφήσει πίσω του μια κληρονομιά σε γερά θεμέλια. Μπορώ να σας πω συμπερασματικά τα εξής Πρώτον, είναι προσιλωμένος και ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του ε, στη δημοκρατία. Και αυτό όχι μόνο για να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει αιτήματα ε, ε, διεθνών θεσμικών οργανισμών ή εξωτερικών. Είναι εσωτερική ζήτηση πρώτα απ' όλα. Ο το ζητάει. Ήταν από τους βασικούς παράγοντες ε, που επέτρεψε να αναλάβει την εξουσία πέρυσι το κόμμα μας, το όνειρο της Γεωργίας. Το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και οικουμενικά και ισχύουν και για την Ευρώπη και για τη Γεωργία. Δεύτερο, η ουσία των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών στη Γεωργία είναι ότι δημιουργούμε θεσμούς δημόσιους, όχι δεν αφορά αυτό άτομα, ας πούμε, πρόσωπα, τον Πρωθυπουργό, υπουργού που ε, προωθούν ε, κάποια ε, μεταρρύθμιση. Δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο θα επιβιώσει και θα ζήσει περισσότερο από οποιοδήποτε πολιτικό και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο. Θεσμοί με διαφάνεια, με εμπιστοσύνη κυρίως των πολιτών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ε, είναι παράλληλη η πορεία μας ταυτόχρονη σε πάρα πολλούς τομείς και πιστέψτε με είναι τεράστια πρόσκληση και τεράστιο έργο αλλά δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Ο λαός της ε, Γεωργίας ε, είναι εταίρος της Ευρώπης. Το ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει από εμά να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή πορεία προς τη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους και παραπέρα ε, και μαζί με σας πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και η σημερινή κυβέρνηση της Γεωργίας είμαι πεπισμένη θα αφήσει ως κληροδότημα μια ευρωπαϊκή πορεία, μια ισχυρή δημοκρατία, θεσμική δημοκρατία που δεν θα μπορέσει καμία ε, μελλοντική γεωργιανή κυβέρνηση να ανατρέψει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Κύριο να καταρχά, το λόγο που έγινε και επικεφαλή αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα. Κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνεργασία με τα κοινοβούλια της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε την Κύριε Υπουργό και να προσθέσουμε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων μαζί της. Ξέρετε ότι καθήκον του Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας είναι να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές ε, συνθήκες για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων κοινοβουλίων των κρατών ε, αυτό έχει προχωρήσει το τελευταίο καιρό ιδιαίτερα μετά τις εκλογές που έγιναν στη Γεωργία πέρυσι, τις οποίες είχα και την ευκαιρία να παρακολουθήσω εγώ. Είχα παραστεί μάλιστα και στην Τυφλίδα, στην οποία επισκέφθηκαν προσωπικό 20 εκλογικά κέντρα όπου μπόρεσα να γίνω μάρτυρας και αυθόρμη των εκδηλώσεων χαράς και ενθουσιασμού για τους ε, νικητές των εκλογών στους δρόμους της πόλεως. Τώρα βλέπουμε λοιπόν μια ειρηνική ε, μετάβαση στην εξουσία και μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας θεσπίστηκε μία κοινή εκδήλωση μεταξύ των δύο κοινοβουλίων μας, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίου της ε, Γεωργίας, μια πρώτη ημερίδα χωρίς ψήφισμα. στην οποία συζητήσαμε και παρακολουθήσαμε ιδιαίτερη ανησυχία την αντιπαράθεση μεταξύ των βουλευτών, της, ε, των κυβερνητικών βουλευτών με αυτούς της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι βεβαίως για περισσότερη συνεργασία, επικοινωνία και καλύτερες ε, σχέσεις και συνεργασία και θα συμβάλλουμε σε αυτό όσο μπορούμε. Πολλοί από εμά και τους συναδέλφους με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουν την ε, ε, επίσκεψη και την παρακολούθηση των εκλογών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την επίσκεψή της και την ειλικρινή τοποθέτηση και περιμένω βεβαίως και τις απαντήσεις της ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, ο εισηγητής μας. Καλώς λέει ο εισηγητής, ο κύριος και ε, Θα μιλήσω και εγώ πολωνικά λοιπόν, αφού μίλησε και ο πρόεδρος αντιπροσωπείας μας τσεχικά. Θα είμαι και πιο ακριβής στα όσα θα πω με τον τρόπο αυτόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της γεωργίας μας έχει απασχολήσει πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο. Μα κάνει πολλές συναντήσεις. Ευχαριστώ την ε, Υπουργό για την ε, ευκαιρία που μας προσφέρει για τα αλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας έδωσε να επισκεφθούμε τον κύριο Χαμπισφίλη στην ε, φυλακή δύο ή τρεις φορές. Χωρίς να υψέρχομαι τώρα σε λεπτομέρειες, θα ήθελα απευθυνόμενος σε εσά ως εκπρόσωπο του κυβερνητικού συνασπισμού να διατυπώσω μια έκκληση προς όλη την κυβέρνηση. Οι προεδρικές εκλογές, οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές πρέπει να υπογραμμίσω έχουν τεράστια σημασία και πιστεύω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους τους πολίτες της Γεωργίας. Θα έχουν τεράστια σημασία λοιπόν οι εκλογές αυτές και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να μετατραπούν σε μια εθνική εορτή, σε, μια μέρα πανηγυρισμού σε ολόκληρη τη χώρα και ελπίζω και εσείς ως κυβέρνηση, ως συνασπισμός κυβερνητικός να συμβάλλετε με όλες σας τις δυνάμεις ώστε να στεφθεί με επιτυχία ε, αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Και ελπίζω, και ήδη από τώρα βέβαια, εν των εκλογών, να προχωρήσετε και να αναλογιστείτε ενδεχόμενο απονομής, ε, ε, κήρυξης αμνηστίας, πολιτικής αμνηστίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζητάω να ανατραπούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες και να αποφυλακιστεί ο, ο επιφανής σας κρατούμενος, αλλά από την άλλη υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ε, ελεχθεί κάποιος είτε με κατοίκον περιορισμό, είτε με δια... άλλα ε, νόμιμα μέσα, κάτι το οποίο πιστεύω θα ήταν προς όφελος και της ε, δημοκρατίας της χώρας σας και Τη εικόνας της σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Αν βρίσκατε μια εναλλακτική ως προς τη φυλάκιση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, πρώτη φορά επισκέφθη τη χώρα σας με την αντιπροσωπεία του κυρίου Ντορζόν τότε, την ε, Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, που είχε ως κύριο μέλημά της βέβαια την ασφάλεια και την άμυνα. Είχαμε την ευκαιρία όμως να συνομιλήσουμε με αρκετούς και με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα τη χώρα σας. Με, το τόσο πλούσιο, με την τόσο πλούσια ιστορία, με τις τόσο σαφείς ε, διασυνδέσεις, με τους τόσο σαφείς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς με μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κατεπλάγει και θα αναφερθώ στους δικούς σας τομείς αρμιδοτήτων, τους ε, Υπουργού Δικαιοσύνης. Γιατί εδώ το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία, η διαφάνεια, ε, η ανώθευτη διεξαγωγή των εκλογών για την επιλογή Προέδρου στη χώρα. Με κατέπληξε λοιπόν το γεγονός ότι διεπίστωσε ότι μπορεί να υπάρχει επιλεκτική ε, δικαιοσύνη. Επισκεφθήμεν τον ε, πρώην Πρωθυπουργό Μαρεμεσβίλη στην φυλακή. Δυόμισι μήνες χωρίς ε, τη δυνατότητα επίσκεψης από τα μέλη της οικογένειάς του είχαν περάσει. Χάρη όμως τη δική μας παρέμβαση και τις δικές σας βεβαίως ενέργειες αντιμετωπίστηκε αυτό. Αλλά πρέπει να πω ότι κατεπλάγει διότι ενώ ήταν σοβαρός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, με την ε, φυλάκισή του και την απαγγελία κατηγοριών, όποιες και είναι αυτές, διαφθορά και το καθεξής, όποιες και είναι αυτές, Και ενώ δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής του στο εξωτερικό, κάποιος δικαστής απεφάσισε και διέταξε την προσωρινή κράτησή του πριν από την δίκη. Δικαστής ο οποίος ο ίδιος είχε καταδικαστεί για διαφθορά όταν ήταν ακόμη υπουργό των εσωτερικών. Αυτό με ανησυχεί βαθύτατα. Ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτή η δίκη το ταχύτερο δυνατό, διότι αυτή η οσμή επιλεκτικής δικαιοσύνης είναι πολύ ανησυχητική και Επίσης ε, το ενδεχόμενο ε, εκλεγμένες τοπικές αρχές ανά την χώρα να υπαχθούν σε έλεγχο, να αμφισβητηθεί δηλαδή το κύρος ήδη διεξαχθήσεων εκλογών και επίσης ε, δηλώσεις από τον αρχηγό της κυβέρνησής σας με εκφράσεις μίσους κατά των ομοφιλοφίλων ή κατά των μη ορθοδόξων που ζουν στη χώρα των μειονοτήτων δηλαδή, ή άλλες τοποθετήσεις σε σχέση με την Ήρμα η βυσβήλει αν δεν απατώμενε το όνομά σας. Το όνομά της. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ανήκουν στο δικό σας πεδίο αρμοδιοτήτων. Είναι όλες οι εξελίξεις πάρα πολύ ενισχυτικές και ελπίζω να έχουν αντιμετωπιστεί πριν την ώρα των εκλογών. Κυρία Νίπλερ έχει το... Νίκολάη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκ μέρους της, ε, της Άλντε για τη Γεωργία αναλαμβάνω εγώ το λόγο. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει ε, νόημα να μιλάμε για ε, μεμονωμένες περιπτώσεις. Εάν ε, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη σε μία χώρα, δεν χρειάζεται να σταθούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η αμεροληψία είναι ύψιστο μέλημα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχω μία μόνο ερώτηση προς εσάς Πώς εκτιμάτε το επίπεδο πολιτικής διαφθοράς στην ε, Γεωργία. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ε, καλωσορίζω και εγώ, λέει η κυρία Λούνατσεκ. Ε. Χαίρομαι που ανταλλάσσουμε πάλι απόψεις μετά την επίσκεψη της ΑΦΕΤ το καλοκαίρι. Σε σχέση με αυτά που προείπαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα κατά Ποιοι να πω αυτά που, αυτό που προείπε και ο κύριος Μπρόκ, ο Πρωθυπουργό ο οποίος ε, απείλησε με παρέτηση μετά την προσχώρηση της Αρμενίας στην ε, Τελωνιακή Ένωση, είπε ο Πρωθυπουργό σας ότι μπορεί να προσχωρήσετε και σας, διότι σας ενδιαφέρει και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, όμως αυτό αποτελεί αντίφαση. Μπορείτε να μας πείτε τι εννοούσε ο Πρωθυπουργό σας, αντανακλά, την ε, θέση της κυβέρνησης για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην υπόθεση Τσέλα αναφερθήκατε σε αυτήν, είπατε ότι η Γεωργία στο μέλλον θα πρέπει να λάβει μία απόφαση για τα κατά πόσο μπορείτε να δεχτείτε τέτοιες ε, μειονότητες ε, στη χώρα σας. Αλλά υπάρχουν και άλλες θρησκευτικέ μειονότητες οι οποίες θα μπορούσαν να μπορέσουν να προσεύχονται όπως θέλουν ε, και να έχουν και ένα μηναρέ στο τζαμί τους. Σε σχέση με τις λεσβίες και τους ομοφιλοφίλους, μας είπα την πρώτη φορά τον ε, Ιούνιο-Ιούλιο ότι όσοι έχουν κατηγορηθεί για βία, δύο από αυτούς ήταν ε, ιερωμένοι, θα συνεχιστεί η δίκη τους. Από όσο γνωρίζω έχουν εγκαταληφθεί αυτές οι κατηγορίες ε, για έλλειψη, λόγω έλλειψη στοιχείων. Αλλά από όσο ξέρω υπήρχαν επαρκή στοιχεία για, την, ε, για κατηγορία. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτές η, αυτή η έκρηξη βίας σε μία διαδήλωση ε, έγινε αποδεκτή. Ναι. Διότι αυτή η ομοφοβία στη χώρα σας στη χώρα σας η ομοφιλοφοβία θα αυξηθεί. Ως προς τον νόμο κατά των διακρίσεων είπατε ότι έχει συνταχθεί, ε, συμπεριλάβατε την κοινωνία των πολιτών όπως προείπατε αλλά φοβούμαστε ότι δεν θα μεταφραστεί ε, στο, σε γράμμα του νόμου πριν από τις εκλογές. Γιατί καρκινοβατεί αυτή η διαδικασία τέλος κάτι σε σχέση με τους ισχυρισμούς ε, στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μυρισβίλη, ο οποίος ε, αυτή τη στιγμή εκτεί την ε, ποινή του. Ναι, τελειώνω, τελειώνω και εσείς μακρηγορήσατε. Από όσο γνωρίζαμε υπήρχαν ισχυρισμοί για ε, ε, κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας. Μπορείτε να μας πείτε τι, ποια είναι τα ευρήματα γύρω από αυτή την υπόθεση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω. Κυρία Υπουργέ, είπατε λέει ο κύριο Σαλαφράνκα, ότι δεν θα κάνετε μία πολιτική δήλωση ή προσέγγιση, αλλά θα ήθελα με βάση τα σχόλια της κυρίας Λούνατσεκ να επεκταθώ κι εγώ και να μας διασαφηνίσετε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δηλαδή τη συμμετοχή στο Ευρωασιατικό πρόγραμμα και σχήμα. Μετά από τις δηλώσεις αυτές, ε, μάλλον πριν από τις δηλώσεις, όπως ξέρετε η Αρμενία είχε προσχωρήσει στην Τελωνιακή Ένωση. Όμως ε, θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ότι πράγματι αυτό ισχύει. Δεύτερον, όπως είμαι και οι προλαλήσαντες και ιδιαίτερα οι φιλελεύθεροι, θα θέλαμε, χωρίς να προδικάσουμε ε, τη θέση του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, πέντε φορές έγιναν δηλώσεις έναντι της εισαγγελικής αρχής, αλλά στη συνέχεια ε, απελευθερώθηκαν οι κατηγορούμενοι. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο πραγματικά υπερασπιζόμαστε και προσπιζόμαστε την εικόνα των ε, υποδίκων και ε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια ελπίζω η διαδικασία του Βίλνιους να στεφθεί από, τη, από επιτυχία και ελπίζω να μου επιβεβαιώσετε το ότι θέλετε να προωθήσετε αυτή τη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μου απαντήσετε σαφώς επί του ερωτήματος αυτού. Um, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις ε, αυτές ευπρόσδεκτες όλες οι ερωτήσεις, διότι όλοι μιλάμε την ίδια ε, ε, τη γλώσσα η οποία μας αρμόζει καλύτερα, γι' αυτό θα συνεχίσω στα γαλλικά. Εγώ προσωπικά, σε σχέση με τα αρχεία που έχουν καταστραφεί, Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν αναλάβαμε την εξουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών ανακαλύψαμε ε, πολλά, πολλές ε, βιντεοτενίες, ε, οπτικοακουστικές και επρόκειτο για υποκλοπές που έγιναν από την Υπηρεσία Συνταγματικής Ασφάλειας. Κύριε Λίζεκ, όπως γνωρίζετε, αυτές οι εγγραφές έγιναν υπό την ε, Πρωθυπουργία Μερασφίλη. Αυτές οι παράνομες ε, εγγραφές, υποκλοπές, χωρίζονται σε δύο τμήματα και ακολουθούμε τις συστάσεις ε, του κυρίου Άμαρμπερ κατά γράμμα. Στο πρώτο τμήμα αυτών των, των βίντεο βλέπουμε ε, προσωπικές στιγμές πολιτικών που βρίσκοντα την αντιπολίτευση τότε και ε, και δείχνουν και την προσωπική ζωή δημοσιογράφων που επέκριναν την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο είναι ότι πρόκειτο για ε, στιγμές της ιδιωτικής ζωής εκείνων που συμμετείχαν στην συμπολίτευση τότε για να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό. Δεν θα ήθελα όμω να μπω σε μια διαδικασία οικοτολογίας. Άρα με τον συνάδελφο, τον Υπουργό Εσωτερικών και τέσσερις εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών πριν από δέκα μέρες καταγράψαμε αυτές τις ε, υποκλοπές και σύμφωνα με τις συστάσεις του κυρίου Αμαρμπέρ τις καταστρέψαμε δημοσία ενώπιον των ΜΜΕ που ε, αναπαρήγαν αυτή την ε, καταστροφή. Η διαδικασία όμως δεν έχει λήξει, διότι υπάρχει ένας ε, εγγενής φόβος στη γεωργιανή κοινωνία, σύμφωνα με τον οποίο ίσως υπάρχουν αντίγραφα που έχουν εξαχθεί από πρώην μέλη της κυβέρνησης που εγκατέλειψε πέρυσι την εξουσία και που έχουν εγκαταλείψει την χώρα πριν από τις εκλογές της 1ης Οκτωβρίου πέρσι για να μην ε, ανακύψουν νέο αυτά τα αντίγραφα και να χρησιμοποιηθούν εκβιαστικά κατά του οποιοδήποτε μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών υποβάλαμε ένα σχέδιο νόμου ενώπιον του Κοινοβουλίου που απαγορεύει την χρήση των παράνομων αυτών αντιτύπων. Μπορεί να υπάρξουν χρηματικές ε, κυρώσεις κατά των υπευθύνων που θα αποτολμούσαν κάτι τέτοιο, αλλά θα θέλαμε οι κυρώσεις να είναι πιο αυστηρές. Δηλαδή, πέρα από τις χρηματικές ε, κυρώσεις να υπάρξουν και σοβαρότερες για να μην ξαναβγούν στην επιφάνεια τέτοια αντίγραφα. Το δεύτερο τμήμα αυτών των ε, υποκλοπών αφορά ε, βασανιστήρια και βιασμούς κατά φυλακισμένων ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. βρήκαμε αυτές τις εγγραφές μέσα σε βαρέλια από που, ε, που ε, γνωρίζουμε για, τα οποία, για τις οποίες υποκλοπές είμαστε σίγουροι ότι ήταν υπεύθυνη η, πρώτη κυβέρνηση, πρώην κυβέρνηση του κυρίου Μερασβίλη. Πρόκειται για εγκλήματα για έγκλημα και θα πρέπει να γίνει η σωστή διαδικασία δίωξης για αυτά, αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Και πάλι ακολουθούμε τις συστάσεις ε, του κυρίου Αμαρμπέρ. Σε σχέση με τις εκλογές, η κυβέρνησή μας καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε στις 27 Οκτωβρίου το βράδυ να παρευρεθούμε στην ε, Εθνική ε, αυτή η νίκη που γνωρίσαν, που γνώρισα και εγώ πέρσι στην ε, πρωτεύουσα πέρσι, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσει αυτή η εμπόλεμη διαδικασία και δεν θα λήξει εάν στις 27 ε, Οκτωβρίου δεν έχουμε διαφανή, μια διαφανή εκλογική διαδικασία που θα επιτρέψει και σε εσά να πείτε ότι διενεργήθηκαν σωστά οι εκλογές με μυστική ψήφο. Ως προς την επιλεκτική δικαιοσύνη, ακούμε πολλά για αυτήν τον τελευταίο καιρό. Εγώ ως πρώην Γενική Εισαγγελέα της χώρας ε, που εγκατέλειψε αυτό το αξίωμα, μπορώ να σας πω ότι όταν αναλάβαμε την εξουσία είδαμε ότι οι, ε, οι εισαγγελικές αρχές της Γεωργίας δεν μπορούσαν να εργαστούν, διότι στο παρελθόν ε, αρκούσε να βρεθείτε ενώπιον ενός δικαστή για να του υπαγορεύσετε την ε, απόφαση. Γιατί ο δικαστής σημεριζόταν τα πάντα. Από τότε που αναλάβαμε την εξουσία, οι γενικοί εισαγγελείς κατανόησαν ότι οι δικαστές αποτελούν μια αυτόνομη αρχή που πρέπει να αποδείξει την ενοχή του οποιοδήποτε. Άρα η μεταρρύθμιση της βασικής εισαγγελικής αρχής συνεχίζεται. Πρόκειται για μια ε, διαδικασία που είναι πολύ πιο ε, δύσκολη ε, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της γενικής, γενικότερα της δικαιοσύνης απέχουμε πολύ από τη βασική αυτή μεταρρύθμιση της εισαγγελική αρχής. Οι δικαστές είναι ελεύθεροι εδώ και δέκα μήνες, αλλά υφίστανται ακόμα ζητήματα και προβλήματα. Με τα δικαστικά μέσα ε, επιτρέψαμε στους δικαστές να δρουν αυτόνομα και αυτόβουλα μέσα στα πλαίσια του, ε, της δικαιοσύνης και να μην εξαρτώνται από τους ιεραρχικά ανώτερους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένας δικαστής δεν αναλαμβάνει μία ε, υπόθεση αυτόματα. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου αποφασίζει ποιος θα ασχοληθεί με τι. Άρα υπάρχουν δικαστές που ασχολούνται με ε, σοβαρές υποθέσεις και άλλους δικαστές που δεν ε, ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις εάν δεν το επιθυμεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές της δικαιοσύνης και χρειαζόμαστε χρόνο έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε το σχέδιο νόμου, διότι κάθε σχέδιο ε, νόμου την χάνει διαπραγμάτευσης ε, με μένα τους υφυπουργού, την κοινωνία των πολιτών και ούτω καθεξής. Ως προς τους μιναρέδες, Υπέστην κριτική από τις δικές μου αρχές ότι ε, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να, δεν θα έπρεπε δεν θα έπρεπε να προβάλλουμε την άποψη ότι θα έπρεπε να αναρτηθεί παραβιάζοντας τον νόμο. Είπα ότι ακόμα κι αν ήταν ε, παράνομη αυτή η οικοδόμηση, αυτή η ανύψωση δεν θα μπορούσαμε να ε, δεχτούμε να κατεδαφιστεί. Εγώ επικρίθηκα γι' αυτό. Δεν υπάρχει πραγματική ανεξιθρησκεία στη χώρα μας. Χρειάζεται όμως ε, διαθρησκευτικός διάλογος διάλογος μεταξύ των θρησκειών και διάλογος μεταξύ κράτους και εκκλησίας και εκπροσώπων των εκκλησιών. Όταν λοιπόν υπάρχουν θέματα ταμπού, βεβαίως ελοχεύει αυτός ο μεγάλος ε, κίνδυνος. Πρόκειται για μία ιστορία που ενόχλησε σε σχέση με τις ε, θρησκευτικές μειονότητες. Δεν θα θέλαμε ε, παρόμοια συμβάντα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για συμβάν, διότι δεν πρόκειται περί αυτού ε, στη γεωργία. Στη γεωργία υπάρχει πραγματική ανεξιθρησκεία. Ως προς την αποχώρηση του Πρωθυπουργού είπα ότι το νέο είναι χειριστό για την κυβέρνηση, αλλά είπαμε ότι χρειάζεται υποστήριξη, υποστήριξη και από πλευράς της ε, κοινωνίας των πολιτών. Ε, θεωρεί ο Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση όπως τον είχε διαβλέψει και οι σχετικές μεταρρυθμίσεις επιτρέπουν, μας επιτρέπουν να πούμε ότι μπορεί να αποχωρήσει μετά από μια διαδικασία ε, διαφάνειας καταπολεμώντας την ε, διαφθόρα πολύ περισσότερο από την προγενέστερη κυβέρνηση και μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία των ε, πολιτών να ανελιχθεί. Η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται μεγάλη βοήθεια. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις μεγάλες μικιό και τίποτα άλλο. Άρα θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να ενισχυθεί για να βοηθήσει την κυβέρνηση στο έργο της, διότι αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του παρελθόντος. Η κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Μερασβίλη δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, δηλαδή να απολογείται στον λαό που την είχε εκλέξει. Ως προς τη Συμφωνία Σύνθεσης θα συνεχίσουμε σε αυτή την οδό, ακολουθώντας αυτή την οδό. Βεβαίως θα συνεχίσουμε αυτή μας την πορεία προσβλέποντας ε, σε αυτή την σύνδεση ως προς την ε, Ευρωασιατική Ένωση αποκλείεται για μας οι Γεωργιανοί έκαναν την επιλογή τους η οποία είναι αμετάκλητη. Δεν πρόκειται όμως μόνο για επιλογές αλλά και για παράλληλες δράσεις. Γι' αυτό το Υπουργείο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε κάθε Υπουργείο εργαζόμαστε σε 24 ώρη βάση έτσι ώστε όπως προαναφέρθηκε στο Βίλνιους αυτή η προσπάθεια να στεφτεί από επιτυχία να φτάσουμε σε μια μεγάλη επιτυχία για τη γεωργία έτσι ώστε να μπορέσουμε και στο δικό μου Υπουργείο να έχουμε χρόνο μεταξύ του Βίλνιους και της υπογραφής για να θέσουμε σε εφαρμογή το ρυθμιστικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει εν μία νυχτή. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα όσο πιο αποδοτικά μπορούμε. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο παρέλειψα κάτι. Εάν ναι, θα ήθελα να μου το υπενθυμίσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Και πιστεύω ειλικρινά ότι η κατεύθυνση που μας δίνεται μας προσφέρει καλές ευκαιρίες να προχωρήσουμε καλύτερα, περισσότερο με το Βίλνιους. Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, πολλές, το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά μπορούμε να εργαστούμε, να αγωνιστούμε στα προβλήματα εκεί που υπάρχουν, όπως ακούστηκε νωρίτερα με την επιλεκτική ε, δικαιοσύνη να συνεργαστούμε και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, αλλά είπατε κι εσείς ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη είναι ένας διαφορετικός αγώνας και μπορεί να προχωρήσει η Γεωργία όπως και η Ουκρανία. Γιατί πάνω απ' όλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών από την εισαγγελία. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και ταυτόχρονα ζήτημα είναι εάν μπορεί ένας ε, δικαστής να εξαρτάται από μία αρχή ε, για, το, για να μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του, για το αν θα ανακληθεί, για το αν θα μετατεθεί. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Εάν θα εξαρτάται ο δικαστής στο έργο του από κάποια άλλη αρχή. Είναι πολύ σοβαρή η δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντική επισήμανση και νομίζω ότι μπορώ εκ μέρους της Επιτροπής να πω ότι ελπίζουμε στο μέλλον ε, να σας ξαναδούμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Τώρα θα ψηφίσουμε. Μία σύσταση της κυρίας Νέιτς. Θέλετε το λόγο. Για μια φορά όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά σε πολυθεύσουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία με την τροποποίηση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την αυτή πλειοψηφία. Τρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Πέντε υπέρ κατά αποχές απερίφθη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ολοκληρώσουμε άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ πέρας 45 υπέρ Μία ψήφος κατά, δύο αποχές εγκρίθηκε. Και συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ τους πάντες.